Συνόδο της Ολομέλειας, ε, οπότε θα μεταβάσω στους αρμοδίους τα ψηφίσματα, δεν βλέπω καμία αντίρρηση και άρα διακόπτεται η Σύνοδος Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας εύχομαι καλό ταξίδι.